Eh, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνούμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξη. Μάλλον πρέπει να έρθουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξη. Πριν όμως να προχωρήσουμε, θα πρέπει για θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Η κυρία Μογκερίνη βρίσκεται σε άλλη αίθουσα, σε άλλη συνεδρίαση. Δεν έχει φτάσει ακόμα εδώ και γι' αυτό παρακαλώ και εσείς να δείξετε λίγη υπομονή.